Και τώρα έχουμε την έκθεση του κύριου Ντράγκητσι. Εκμάθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο. Ο εισηγητής, τέσσερα λεπτά. Mr. Chairman, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο παρόν, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Ευρωπαρόμετρο του 2014, το 71% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι δεν είναι πολύ καλά πληροφορημένο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 44% θεωρεί ότι έχει περιορισμένη γνώση για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 52% θεωρεί ότι η φωνή τους δεν προσμετράται. Και γι' αυτό δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι οι πολίτες θεωρούν ότι είναι πολύ μακριά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι ευρωσκεπτικιστές και λαμβάνουν υπόψη μόνο το δημοκρατικό έλλειμμα εκεί που υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε το διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία μας και σε άλλους θεσμούς έτσι ώστε να πληρωθεί το μεγάλο χάσμα που υπήρχε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών και για να αποκατασταθεί, η εμπιστοσύνη τους στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό είναι όλο ένα και πιο σημαντικό μέσα στα πλαίσια της προσφυγικής κρίσης και των σοβαρών απειλών κατά της ανθρώπινης ζωής λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών. Γι' αυτό θα πρέπει ήδη από το σχολείο να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες μέσα στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής ολοκληρωμένης Ευρώπης και έτσι όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργεί και το ότι αποτελεί φυσικά προστιθέμενη αξία. Θα ήταν μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πώς επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χώρα τους και τις δραστηριότητες τους. Έτσι θα μπορέσαν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα θα οδηγούσε σε έναν μεγάλο διαφρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο και γι' αυτό ακριβώς ε, θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ορατή στα, στη διδακτέα ύλη και εκτός διδακτέας ύλης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαβίου μάθηση βεβαίως. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο και των κρατών μελών στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να τονίσω το θέμα της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην διδασκαλία της ιστορίας, για να γνωρίζει κανείς πώς ε, λειτουργήσε το παρελθόν και πώς ε, μπορεί να επιδράσει στο παρόν. Έτσι, μέσα στα πλαίσια αυτής της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, θα μπορούσαν ε, οι ενεργοί πολίτες να μπορέσουν να εισακουστούν σε πλουραλιστικές κοινωνίες. Θα πρέπει να υπάρχει ανεξιθρησκεία και ανοχή. Μέχρι τώρα η πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν ε, εντάξει στη διδακτέα ύλη και τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν πολλά χάσματα μεταξύ κρατών μελών. Ως προς τη διδακτέα ύλη θεωρούμε ότι τα μαθήματα και η διδακτική μέθοδος θα μπορούσε να αλλάξει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα σε, και σε όλα τα φόρα εκτός ε, σχολείου. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν μαθητές πολύ περισσότερα ε, και πολύ καλύτερα ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά την, ε, διαδικασία διδασκαλίας αλλά και, εκτός, και προγράμματα εκτός σχολείου. Αυτό θα βοηθούσε και τους διδάσκοντες και τους μαθητές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα που υπάρχουν για διαπολιτισμική κατανόηση, και για ολοκλήρωση γνώσεων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρηματοδοτική ενίσχυση και θα πρέπει να τονίσουμε και το θέμα της κινητικότητας για τους διδάσκοντες έτσι ώστε και οι μειονεκτικές ομάδες να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ανταλλαγή διδακτικής ύλης ενδοκινοτικά μέσα στα πλαίσια της ε, ε, εκπαίδευσης των πολιτών. Θα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη αυτή τη νέα διάσταση της εκπαίδευσης και μέσα στα πλαίσια ενός κοινού πλαισίου γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να είναι ενεργοί πολίτες ε, οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστώ πολύ και τους Κιώδης. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Μου μένουν πέντε λεπτά για το Καρστιάι. 18 συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Παρακαλώ να δείξετε και εσείς κατανόηση αν δεν μπορούσα να δώσω το λόγο στους ε, πάντες. Πρώτος, πρώτη η κυρία Κομοντίνη Καρσίου. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίσουμε την ευρωπαϊκή ε, ποικιλότητα που υπάρχει και επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρίζος παστικοποίησης θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τις ευρωπαϊκές αυτές αξίες. Οι νέοι μας θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού οι φοιτητέ θέλουν να κατακτήσουν την Ευρώπη, να την οικειοποιηθούν. και αυτό θα πρέπει και ο να λάβουμε υπόψη ότι ο πολιτισμός και οι αξίες κινούνται πέρα από τη διδακτέα ύλη. Θα πρέπει και οι διδάσκοντες να έχουν τα κατάλληλα μέσα και θα πρέπει να υπάρχει και συνεχής κατάρτιση για τους δασκάλους και τους καθηγητές μέσα στα πλαίσια της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, μέσα στα πλαίσια και του e-learning. Ευχαριστώ. Η κυρία λέει ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, η εκπαίδευση είναι η βάση της κοινωνίας και θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα της ευρωπαϊκής ε, διάστασης είναι πολύ σημαντικό ε, μέσα στα πλαίσια γενικότερα της ε, μάθησης, της μαθησιακής διαδικασίας στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και στον τεχνολογικό τομέα και θα πρέπει να συνεχίσουμε και με την επαγγελματική κατάρτιση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το, ο, ο αγροτικός τομέας επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να αποτελέσει σημαντική συνιστόσα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Κιτσίκ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλοί είναι οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις ε, για τις βάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια και τα θεσμικά της όργανα και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η δράση στις χώρες τους. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιληφθεί ο πολίτης πώς ευεργετεί τον καθημερινό του βίου Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμεί να του δείξουμε καθημερινά τι κάνει για τον καθένα μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσουμε το διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία μα, στι ενώσει πολιτών, στου δημόσιου φορεί. Ιδιαίτερα με δεδομένη τώρα της, ε, την κατάσταση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό είναι απαραίτητο. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη τη, Πρέπει να καταστεί σαφές για τον κάθε πολίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εγχείρημα κοινό των κρατών μελών. Κοινή ιστορία και διαφορετικού πολιτισμού εκφράζει. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η ενσωμάτωση λοιπόν τη εκμάθηση στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η εκπαίδευση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει σημασία αρκεί να μην γίνεται μονομερής προπαγάνδα προς τους μαθητές. Πρέπει να κοιτάμε ποιες είναι, ποιες είναι οι πραγματικές προοπτικές της Ευρώπης, αλλά εδώ δυστυχώς η έκθεση δεν αντικατοπίζει την πραγματικότητα. Και λέω ότι μπορεί η απουσία εκμάθησης να οδηγεί σε δημοκρατικό έλλειμμα και ε, ευροσκεπτικισμό. Κοιτάξτε, το δημοκρατικό έλλειμμα δεν είναι συνέστημα, είναι γεγονός και ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι κάποια αρρώστια, αλλά μια γενική ε, συμπίληση τάσεων που δεν εστιάζονται στην Ένωση ως παραγοντέρα του μέλλον. Στόχος είναι λοιπόν ο μαθητής να ετοιμάζεται για μια υφιστάμενη όντως πολυπολιτισμική κοινωνία, πρέπει ωστόσο να ενισχυθεί η ταυτότητα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μια ταυτότητα η οποία χάνεται όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, Αντινόλφη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει οι πολίτες για να αισθανθούν Ευρωπαίοι να γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να διαθέτουν όλα τα μέσα υλικά και πνευματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρχει μία κριτική σκέψη σε σχέση με την ευρωπαϊκή ιστορία και να προωθήσουμε επίσης τα κοινά θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιπτώσει στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν θα υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Το δημοκρατικό έλλειμμα αναγνωρίζεται και από την ίδια την έκθεση και τονίζεται ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα πρέπει να επανορθωθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποκτάν Βέντα, τελευταίος στη διαδικασία Καστία. Ένα λεπτό. Πρόεδρε... Πρόεδρε, Είμαι υπέρ της εισαγωγής ε, ε, τέτοιου μαθήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην σχολική ύλη, γιατί η γνώση αυτών των ζητημάτων, αλλά και του αντικτύπου της ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, μπορεί να αποτελέσει τμήμα ευρύτερων κοινωνικών γνώσεων που θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μαθητής. Είναι λοιπόν μια προσταθεμένη αξία και εφοδιάζει τους ε, μαθητές με απαραίτητες ε, γνώσεις ε, για τη σημερινή πραγματικότητα. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει και ευρύτερη διαπαιδαγώγηση, όχι μόνο με την εκμάθηση αυτών των μαθημάτων. Λαμβάνοντα υπόψη τώρα και την εισρωή μεταναστών και το πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε πλέον, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μνήμα σε ό,τι αφορά και την ε, ε, ένταξη αυτών των μεταναστών στην κοινωνία μας. Το αναφέρει και ο εισηγητής αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τώρα εκ μέρους Επιτροπής ο κύριος Ναύρατσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε ξέρετε κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση για την εκμάθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον κύριο Ντράγκη για την ε, εξαίρετη δουλειά του. Τελευταίε εκθέσει έχουν δείξει, δείξει για άλλη μια φορά τον κίνδυνο του ε, να αποκοπεί ο νέο ε, από το ενδιαφέρον του για την ε, κοινωνία. Μια τέτοια εκπάθηση λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύπλευρη και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης. Κάθε νέος στην Ευρώπη πρέπει να αντιλαμβάνεται και να συμμερίζεται τις θεμελιώδες μας αξίες. Πρέπει να χτίσουμε μια Ευρώπη όπου κάθε νέος θα μπορεί να βρει τη θέση του στην κοινωνία και να αναπτύξει το δυναμικό του δεδομένου του περιβάλλοντος από το οποίο προέρχεται και των ικανοτήτων του βεβαίω. Τι σημαίνει αυτό τώρα η εκμάθηση Ευρωπαϊκής Ένωση στο σχολείο. Γενικά συμφωνώ με την προσέγγιση του κ. Ντρακίτση στην έκθεσή του. Για μένα έχει να κάνει με δύο κύριες πτυχές. Την διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας, των πολιτισμών, των γλωσσών αφενός και ε, αγωγή του πολίτη αφετέρου. Εδώ όντω έχουμε να κάνουμε με δύο αλληλένδετε πτυχέ. Αν δεν γνωρίζουμε την Ευρώπη, είναι αδύνατο να αντιληφθούμε τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, όταν μαθαίνει κανείς τις γλώσσες και το, η κουλτούρα των γειτόνων του, ε, ενισχύεται και η αίσθηση τη ηθαγένεια. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ε, ενσωμάτωση της εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως ζητάει ο κύριος Τραγκίτσι. Βεβαίως τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ενσωματώσουν στα εθνικά προγράμματα σπουδών τους τα ε, ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ γίνεται λόγος εκ μέρους του ΣΥΓΙΤΟΥ μόνο για συνεργασία με το των μελών και ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος Erasmus Plus. Πριν από μερικά χρόνια το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο συμφώνησε στην ένα βασικό σύνολο γνώσεων που θα πρέπει να έχει κάθε ε, πολίτης δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο και θα διευκολύνει το νέο μας να γίνει υπεύθυνο πολίτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι απαραίτητο περισσότερο τώρα από ό,τι ποτέ να καταλάβουμε καλύτερα αλλά πάνω απ' όλα να να μεταγγίσουμε καλύτερα τις ε, αξίες μας. Το Μάρτιο του 2015, πριν από ένα χρόνο, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εκπαίδευση με τη διακήρυξη των Παρισίων ε, έδωσαν την απάντησή τους μετά τις επιθέσεις του Σαρλί Εμπτό για την αγωγή του πολίτη, για την προαγωγή των αξιών της ε, διαλλακτικότητα, της αποτροπή των διακρίσεων και στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 έχουμε ενσωματώσει τέτοιες ιδέες στις συνεργασίες με τα κράτη-μέλη. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την βία ριζοσπαστικοποίηση, την ενίσχυση της ε, κριτικής σκέψης ε, και την ε, επαγνύπτυνση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η σημασία που αποδίδει έκθεση στο Erasmus Plus, στο Europe for Citizens, στο Creating Europe, τέτοια προγράμματα ευρωπαϊκά που ενθαρρύνουν και την υπαγένεια και την εκμάθηση των γλωσσών και την ε, ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πρόγραμμα του 2016 παραμένει ε, ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται τα προγράμματα αυτά τα οποία ενθαρρύνουν ε, την αγωγή του πολίτη, τον ενεργό Ευρωπαίο πολίτη. Με το e-twinning, με το δίκτυο 300.000 δασκάλων, με συστήματα που προβάλλουν πλατφόρμες δασκαλίας ηλεκτρονικές στην Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε πολλά για τους δασκάλους μας, για τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει κέριο ρόλο. Έχουμε να κάνουμε πλατφόρμες λοιπόν οι οποίες εξασφαλίζουν ε, διδακτικό, προσωπικό, διδακτικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και επιτρέπουν την ε, ανταλλαγή των πρακτικών. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του ε, της την αξιοποίηση αυτών των μέτρων και την ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των πολιτών που προκύπτει από αυτά. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερω λοιπόν και για την ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων στην κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, προσβλέπω σε περαιτέρω συνομιλίες μαζί για τα θέματα αυτά. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση.